Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στη σημερινή μας συνεδρίαση. Δεν είμαστε ακόμη πολύ άριθμοι, αλλά ελπίζω ότι θα φτάσουν και άλλοι στο μεταξύ. Η επόμενη μας κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΜΠΛ και ΦΑΜ είναι στις 12 Ιουλίου. Εκεί θα εγκρίνουμε και την έκθεση. Την έκθεση δηλαδή που θα συζητήσουμε σήμερα σε αυτήν την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης και ε, Δικαιωμάτων της Γυναίκας. Τούτου λεχθέντος, ας περάσουμε στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης που προβλέπει την δημιουργία προϋποθέσεων στην αγορά εργασίας ε, που θα ευνοούν το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπλινκεβιτσούτη που είναι η συγγήτρια από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη συνάδελφος Δάνοκα για τη βοήθειά της και να ευχαριστήσω και τους και οδησηγητές, καθώς και τους υπόλοιπους συναδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίες. Οι τροπολογίες έδειξαν ότι όλοι μας προβληματιζόμαστε από την επιδείνωση της δημοκρατικής κατάστασης στην Ευρώπη και να γνωρίζουμε την ε, επιτακτική ανάγκη αναζήτησης λύσεων για να αυξήσουμε τη γεννητικότητα Ταυτόχρονα θα πρέπει να παράσχουμε φροντίδα σε παιδιά, σε εξαρτημένους, δηλαδή ηλικιωμένου ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρίες. Επίσης, ε, συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να, να μπορεί να συνδυάζει κανείς την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή και να υπάρχει μια πιο ακριβωδή και κατανομή των υποχρεώσεων και των ευθυνών ε, ε, μεταξύ των μέλων της οικογένειας και μεταξύ των δύο φίλων κυρίως. Βέβαια, ω προ το στόχο συμφωνούμε, αλλά ω προ το μέσο και τα μέτρα για να το επιτύχουμε έχουμε μερικέ διαφορέ μεταξύ των ε, πολιτικών ομάδων. Άλλοι είναι υπέρ ε, νομοθετικών μέτρων, άλλοι υπέρ πιο λιγότερο δεσμευτικών προαιρετικών μέτρων ή συστάσεων. Πάντως, δεδομένου ότι ο στόχος μας είναι κοινό, ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάντως επανειλημμένως διαβεβαίωσαν την Επιτροπή μας ότι μέχρι τα τέλη του έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει μια δέσμη νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων με αντικείμενο το συνδυασμό του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου. Εμείς στις δύο επιτροπές ε, θα αναζητήσουμε συμβαστικές λύσεις που θα περιλαμβάνουν και νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα. Πάντως προσωπικά χαίρομαι ιδιαίτερος για το μεγάλο αριθμό των τροπολογιών που τάσσονται υπέρ της μεταποδοχών ε, άδειας πατρότητας και μάλιστα τα πλήρους αμοιβή. Έτσι θα μπορέσουμε να κατανείμουμε πιο ισότιμα τις οικογενειακές υποχρεώσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών με τέτοια αμοιβόμενη, πλήρως αμοιβόμενη άδεια πατρότητας. Και θα ενισχύσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, ώστε να μπορούν να έχουν μια σταδιοδρομία πιο απρόσκοπτη. Επίσης θα πρέπει να σεβαστούμε τους στόχους της Βαρκελόνης, δηλαδή να βελτιώσουμε την, την πρόσβαση σε ποιοτικέ και ε, από προσιτές ως προς την ποιότητα και την τιμή υπηρεσίες παροχής φοροντίδας για τα παιδιά. Έχουμε επίσης κάποιες τροπολογίες που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα των ανάπηρων παιδιών. Γιατί όλοι γνωρίζουμε από την άλλη ότι ο πληθυσμός μας γυράσκει, ενώ το προσδόκιμα της ζωής αυξάνεται. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Έχουμε πολύ καλές τροπολογίες για τη φροντίδα ηλικιωμένων, για τις επενδύσεις σε πιο μακροπρόθεσμες υπηρεσίες φροντίδας, που επίσης θα πρέπει να είναι προσιτή και σε σχετικά χαμηλές τιμές. Και επίσης θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη και τις ε, δυνατότητες άδεια για τους παρέχοντες φροντίδα. Υπάρχουν σχετικές τροπολογίες. Διαπιστώνουμε ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι σχετικά χαμηλή σε σχέση με αυτή των ανδρών. Γι' αυτό στην έκθεσή μου απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την επαναφορά, επιστροφή των γυναικών στην αγορά εργασίας και τις προϋποθέσεις ε, για τους άντρες να αναλάβουν και αυτοί ένα μεγαλύτερο τμήμα των οικογενειακών ευθυνών και υποχρεώσεων. Έτσι θα εξασφαλίσουμε ισότητα ευκαιριών και στην αγορά εργασίας για τα δύο φύλλα. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα ενιαίο μοντέλο για τη συμφιλίωση στον συνδυασμό επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. Θέλουμε μοντέλο που να ανταποκρίνεται στις ατομικές μας ανάγκες για να μπορεί ο καθένας να συνδυάσει την οικογενειακή με την επαγγελματική του ζωή και να αναζητήσουμε τις λύσεις σε διαφορετικά επίπεδα και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό. Επίσης οι εργοδότες θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτοι στις ε, εργασιακές συνθήκες και θα πρέπει αυτές οι εργασιακές συνθήκες να είναι φιλικές προς τον εργαζόμενο. Χθε είχαμε δύο συναντήσεις με τους και ηγητές ε, των δύο επιτροπών Τρίτη και Πέμπτη και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συνενετικές λύσεις. Εγώ ως εισηγήτρια της Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων της Γυναίκας ε, επικεντρώθηκε κυρίως σε θέματα ισότητας ε, των δύο φύλων, ενώ η συνάδελφος η Τατιάνα Σδάνοκα, που είναι η αρμόδια εισηγήτρια, είναι εισηγήτρια από την Επιτροπή Απασχόλησης, θα επικεντρωθεί στο θέμα που άφηνε περισσότερο των αρμοδιοτήτων και των ενδιαφερόντων της Επιτροπής Απασχόλησης. Ευχαριστώ. Κυρία Σδάνοκα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την συνεισηγήτριά μου, την κυρία Μπλικεβιτσούτε και τους και ηγητές, καθώς και τους βοηθούς μας, τους συμβούλους μας, το επιτελείο μας, γιατί όλοι συνεργαστήκαμε πολύ επικοδομητικά και καταλήγουμε σε κοινέ λύσει. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε η προλαλήσασα. Πριν περάσω σε πιο ειδικά θέματα που αφορούν την Επιτροπή Απασχόληση, θα ήθελα να επισημάνω ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε. Ε, όταν λάβαμε τις τροπολογίες για το γενικό, το εισαγωγικό τρίμα της έκθεσης που είναι πιο ενιολογικό και επίσης τροπολογίες για τον τίτλο της έκθεσης. Φυσικά δεν μπόρεσα να ελέγξω τους τίτλους και στις 23 μεταφράσεις. Στις ε, γλώσσες πάντως που εγώ γνωρίζω διαπίστωσα ότι υπάρχει κάποια παρεξήγηση με τους τίτλους στα, στο πρωτότυπο που είναι αγγλικά μιλάμε για work-life ε, balance, δηλαδή για την ισορροπία μεταξύ εργασίας ε, και ιδιωτικού βίου. Στα λετωνικά δεν είναι ακριβώς ε, η ίδια η μετάφραση. Και στα γερμανικά επίσης λέμε κάτι παρεμφερές, αλλά όχι ακριβώς το ίδιο. Και στο πρώτο τμήμα του γενικού σκέλους, στο πρώτο του Γενικού Τμήματος της έκθεσης, επισημαίνουμε ότι ο συνδυασμός της επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής θα πρέπει να εξασφαλίζεται ως θεμελιώδης δικαίωμα όλων των ανθρώπων. Ε, κατατέθηκαν τροπολογίες που από τις τρεις αυτές λέξεις ε, κρατάνε μόνο τη τις δύο. Μερικές πολιτικές ομάδες δεν θέλουν να φέρεται οικογενειακός βίος, family life. Άλλες ομάδες δεν θέλουν να περιλαμβάνει το ιδιωτικός βίος, private life. Ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία τελικά και θα κρατήσουμε και τις τρεις λέξεις, ώστε να έχουμε τη διαφοροποίηση μεταξύ οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Ε, οικογενειακού συγγνώμη, και ιδιωτικού βίου. Γιατί μιλούμε για διαφορετικέ πτυχέ τη ανθρώπινη ζωή. Άλλο οικογενειακό, άλλο ιδιωτικό βίο. Δεν ταυτίζονται ακριβώ αυτοί οι όροι. Οπότε δεν μπορούμε να αφαιρούμε μερικές λέξει και να κρατούμε μόνο άλλε. Εδώ έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, γιατί πολλές τροπολογίες ε, αφορούν αυτό ακριβώς στο γενικό τμήμα παραγράφους 1 και 6 με τη διαφοροποίηση αυτών των τριών πτυχών που άλλοι τις κάνουν δύο και θα ήθελα οι σκιώδεις ηγητές ε, να μου πούν τη γνώμη τους ποιος ο λόγος που κατέθεσαν αυτές τις τροπολογίες και δεν ξέρω τι, να, τι θα κάνουμε. Ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την ε, διερμηνία για να αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις με τους τίτλους και τις διατυπώσεις. θα ήθελα να διαπιστώσω μία διαφορά στις προσεγγίσεις που έχουμε σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές προτάσεις. Καταρχήν, για το θέμα της άδειας πατρότητας και τη σχετική οδηγία. Και εδώ έχουμε διάσταση απόψεων και μερικές φορές και αντιφατικές, αντιμαχόμενες ε, αποφάσεις ό,τι αφορά την ελάχιστη υποχρεωτική και μη μεταβιβάσιμη άδεια μεταποδοχών για τους πατέρες. Εδώ η Επιτροπή των Δικαιωμάτων της Γυναίκας ίσως έχει διαφορετική γνώμη. Διαπιστώνω βλέποντας και τις τροπολογίες από την Επιτροπή Γυναικών. Εγώ θα προτείνω μια εξορρόπηση της διάστασης απόψεων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση, την ίδια λύση για όλες τις οικογένειες και για όλα τα κρατημέλη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις παραδόσεις, και δεν μπορούμε να επιβάλλουμε μια δεσμευτική διάταξη σε ένα τόσο λεπτό θέμα που είναι η οικογενειακή ζωή και ο επιμερισμός των ευθυνών και υποχρεώσεων εντός μιας οικογένειας. Εμείς ως Επιτροπή Απασχόλησης θα θέλαμε να τονίσουμε όχι μόνο το θέμα των φίλων, αλλά να μιλήσουμε για αυτούς που παρέχουν φροντίδα. Και θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη ε, μιας οδηγίας για τις άδειες αυτών των ατόμων που παρέχουν φροντίδα. Και εδώ υπάρχει διαφορά μεταξύ των κρατών Άλλα είναι πολύ προηγμένα στη σχετική νομοθεσία που καλύπτει τέτοιου είδους ζητήματα και άλλα υστερούν και αφήνει το θέμα της παροχής φροντίδας, αφήνει το θέμα της παροχής φροντίδας ε, στην ιδιωτική σφαίρα. Χωρίς καμία ρύθμιση αφήνει το ζήτημα στην κάθε οικογένεια. Με γνωστές κοινωνικές συνέπειες και ανύπαρκτη σχεδόν κοινωνική προστασία για τους παρέχοντες φροντίδα. Οπότε προτιμώ να βάλω τελεία εδώ και να ακούσω τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών. Και άμα επιτρέπετε θα μιλήσω εκτενέστερα στη δευτερολογία μου. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ζανόκα. Κοιτάξτε για το γλωσσικό. Θα ήθελα να επανέλθουμε στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί και μετά θα ακολουθήσει πολιτική συζήτηση διότι είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις από αυτού. Η διατύπωση που χρησιμοποιεί κανεί στην πολιτική λέει πάρα πολλά και για το περιεχόμενο ενός θέματος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα το λύσουμε σήμερα το θέμα αυτό εδώ. Και τώρα θα μου επιτρέψετε να παραδώσω ε, για λίγο την Προεδρία στην Πρόεδρο της Επιτροπής ε, Γυναικών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Όλσκοκ και καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα δώσω το λόγο τώρα στους και συγγητές των πολιτικών ομάδων. Αφού ακούσαμε τις παρουσιάσεις από τις συνεισηγήτριες των Επιτροπών Γυναικών και Απασχόλησης, για το θέμα του τίτλου, το πρόβλημα δεν είναι γλωσσικό, ο τίτλος είναι σαφής. Μιλά για ιδιωτική ζωή, όχι οικογενειακή ζωή. Άλλο τώρα να πω πολιτική άποψη, κάποιοι βουλευτές θέλουν να το αλλάξουν και να βάλουν οικογενειακή ζωή αντί ιδιωτική. Αποδεκτή και εύλογη θέση τους, αλλά είναι πολιτική αυτή η στάση και όχι γλωσσική. Ο τίτλο είναι προσδιορισμένο και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίτλο έκθεση πρωτοβουλία γιατί έχει εγκριθεί από τη διάσκεψη των Προέδρων. Και ο τίτλος τη Έκθεση είναι αυτός που αναφέρεται στα αγγλικά που μιλά για συνδυασμό επαγγελματική και ιδιωτική ζωής και όχι οικογενειακής. Τώρα, αν κάποιοι ευρωβουλευτέ θέλουν να μιλήσουν και για τι συμφιλίωση με την οικογενειακή ζωή, έχουν απόλυτο δικαίωμα να καταθέσουν σχετικές τροπολογίες. Πάντως επαναλαμβάνω, ο τίτλος της έκθεσης πρωτοβουλίας που θα μείνει αμετάβλητος γιατί έτσι έχει εγκριθεί είναι ο συνδυασμός της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Θα δώσω τώρα το λόγο στο Σκιώδη εισηγητή του ΕΛΚ, τον κύριο Πλούρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω την άποψη του κυρίου Ξίστοφ Χέιτμαν, που είναι ο σκιώδης ηγητής της έκθεσης, αλλά δυστυχώς κολλείται σήμερα και τον αναπληρώνω εγώ, κυρίες και κύριοι. Και η έκθεση, αλλά και η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών δείχνει ότι το θέμα αυτό του συνδυασμού επαγγελματικής και δυτική ζωής είναι πολύ περίπλοκο. Γι' αυτό και θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια σφαιρική προσέγγιση στο ζήτημα αυτό, μια πιο ολιστική προσέγγιση. Πολλέ χώρε ε, μέλη, αλλά και πολλοί ευρωβουλευτέ, ε, επισήμαναν το ζήτημα, το, το ζήτημα της φροντίδας των παιδιών και του επιμερισμού των ευθυνών ε, μεταξύ και των δύο γονέων. Και εγώ πιστεύω ότι το θέμα του επιμερισμού των ευθυνών τη φροντίδα των παιδιών είναι πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει να δημιουργήσουμε προποθέσει ώστε και οι δύο γονεί να μπορούν ελεύθερα και με ίσους όρους να λάβουν γονική άδεια μεταποδοχών. Επίσης είναι πολύ σημαντική η δημιουργία πρόσβασης σε καλής ποιότητας ε, υπηρεσίες ε, φροντίδας παιδιών ε, σε προσχολική ηλικία, δερφονιπιακή σταθμή, παιδική σταθμή και ούτω καθεξής. Γιατί συμφωνώ ότι κάποιες άτυπες μορφές εργασίας ή χαμηλές αμοιβέ η αβεβαιότητα στην απασχόληση είναι όροι που δυσκολεύουν τον επαγγελματικό βίο των γονιών. Και ίσως ε, μερικοί γονείς, κυρίως ε, που έχουν τέτοια προβλήματα, προτιμούν να μην κάνουν καν παιδιά για να αποφύγουν αυτές τις δυσκολίε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις δημογραφικές προκλήσεις και το χαμηλό βαθμό γεννητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, συμφωνώ ότι το θέμα της ισορροπίας, ε, του συνδυασμού μεταξύ ε, επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στο ζήτημα τη φροντίδα των παιδιών. Κάθε πολίτη τη Ένωση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζει ε, τη ζωή του, όχι μόνο στον εργασιακό χώρο, αλλά και στην οικογένειά του, στην αναψυχή, στην ε, προσωπική του ανάπτυξη ή στις συναντήσεις με φίλους. Έχουμε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε στον τομέα αυτό λοιπόν και ίσως θα πρέπει να ρυθμίσουμε και το ζήτημα του ωραρίου εργασίας, ε, το θέμα της προστασίας από απολύσεις, κυρίως των γυναικών και επίσης ε, σωστή κατάρτιση, επαγγελματική και διαβίω εκμάθηση. Επίσης, καλό θα ήταν στην έκθεση αυτή να μην επικεντρωθούμε μόνο στις υφιστάμενες απειλές, αλλά να τονίσουμε και τις ευκαιρίες, το δυναμικό που υπάρχει από μια τέτοια κατάσταση. Και κυρίως να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η εξ αποστάσεως εργασία, η εργασία κατοίκων. Είναι πολύ σημαντικές δυνατότητες. Πολλές τροπολογίες κατατέθηκα για την έκθεση, πολύ αξιόλογες και ελπίζω ότι θα ληφθούν υπόψη από τις δύο συνεισηγήτριες κατά την κατάρτιση συμβαστικών τροπολογιών. Βέβαια, μερικές τροπολογίες είναι παρατραβηγμένες. Ε, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι χρειαζόμαστε φιλόδοξες μεν ε, προτάσεις, αλλά να αποφύγουμε πολύ υπερβολικό προστατευτισμό και μεγάλη επέμβαση είτε στην αγορά είτε στις ε, αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών μελών. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι για πολλά θέματα, κυρίως με νομική ισχύ, θα πρέπει να φροντίσουμε ότι οι φυστάμενες διτάξεις πρώτα απ' όλα θα πρέπει να τηρηθούν πριν περάσουμε στη θέσπιση νέων νομοθετικών διατάξεων. Ελπίζω πάντως ότι και στη συνέχεια των εργασιών θα συμβάλλουμε όλοι στην διαμόρφωση μιας καλής έκθεσης που είναι πολύ σημαντική και περίπλοκη. Ευχαριστώ. Ε, thank you. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, ξεκινάμε τον κατάλογο των ε, ερωτώντων και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκάλπελτς. Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ως σκιώδης ηγήτρια του ΕΛΚ να πω ότι η έκθεση είναι πολύ σημαντική. Και εγώ στηρίζω ε, την ισορροπία που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή. Αυτή είναι πρώτη προτεραιότητα για το ΕΛΚ. Και με μεγάλη χαρά άκουσα αυτά που μας είπε η συγγήτρια, συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Επίσης ε, θέλω να σας πω ότι πρέπει να ζητήσουμε συμβαστικές προτάσεις, γιατί το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει λοιπόν η οικονομική κρίση και επιπρόσθετα υπάρχει και η δημογραφική κρίση στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως ε, μπορείτε να δείτε και στις τροπολογίες που έχω καταθέσει εγώ και οι συνάδελφοί μου στην ε, αγορά εργασίας ε, πολύ συχνά συμβαίνει το εξής. Υπάρχουν ε, ανελαστικές συνθήκες εργασίας, ε, περίεργα ε, ωράρια εργασίας και, και αυτό είναι το πρόβλημα που δεν υπάρχει ισορροπία. Επίσης, ε, δεν είναι ικανοποιητική η κινητικότητα. Είναι πολύ ακριβό το να μετακινείται κανείς και υπάρχει και έλλειψη παιδικών σταθμών, βρεφονιπιακών σταθμών δεν υπάρχει επάρκεια πόρων που να ε, χορηγούνται σε οικογένειες και σε μεμονωμένα άτομα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρόκειται για μία αυτοτροφοδοτούμενη ένταξη, ένταση και συνεχίζεται η ανισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή. Οφείλουμε λοιπόν να ρίξουμε φως ε, στο πρόβλημα και εγώ συμφωνώ με το συνάδελφο από το ΕΛΚ που ανέφερε ότι ο πρωταρχικός μας στόχος δεν είναι να θεσπίζουμε συνεχώς ε, νομοθετικές διατάξεις, ενώ δεν μας ενδιαφέρει η εφαρμογή των ήδη, ιστα... Ε, ε, υφιστάμενων. Πρέπει να αναζητήσουμε τα αίτια του προβλήματος, όπως επίσης και την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων. Ε, προφανώς και υπάρχουν στα 28 κρατημέλη διαφορετικές ε, νοοτροπίες, διαφορετικές νομοθετικές διατάξεις. Εμείς οι γυναίκες αντιμετωπίζουμε διαφορετικά όλα αυτά τα προβλήματα. Προφανώς και δεν υπάρχει ένα μοντέλο που να βολεύει όλους. Ε, το πρόβλημα ποικίλει ανάμεσα στα κρατημέλη και στην προσέγγιση του καθενός για το ποια είναι η σωστή λύση. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε αυτό το θέμα κατά νου και δεν πρέπει να επιβάλλουμε ένα ε, μοντέλο εκ των άνω προς τα κάτω. Ε, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε οτιδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό. Θέλω να ελπίζω ότι την επόμενη Τρίτη και την Τετάρτη θα βρούμε συμβαστικές προτάσεις στη συνεδρίαση των σκιωδών. Και επίσης ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας και να μεριμνήσουμε και για τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις. Όλα αυτά τα θέματα είναι εθνικής δικαιοδοσίας, άρα η λύση μπορεί να βρεθεί ε, πάνω απ' όλα σε εθνικό επίπεδο, βέβαια με κοινούς στόχους και αυτοί οι κοινοί στόχοι πρέπει όμως να ε, διευκρινιστούν σε αυτή την έκθεση και να ε, ορίζονται και ξεκάθαρα από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε κυρία Γκαλπέλτς εκ μέλου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών. Το λόγο έχει η κυρία Τζεντήλε από την Επιτροπή Απασχόληση. Ευχαριστώ πολύ και τις ε, δύο Προέδρους. Έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση όσο έχει διαμορφωθεί ε, θα πρέπει ε, το όλο θέμα να το επανεξετάσουμε γιατί υπάρχουν ε, διαφορετικές προσεγγίσεις και οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις οφείλονται και στο ότι κάθε κράτος μέλος έχει κάνει και διαφορετικές εμπειρίες. Όσον αφορά τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, νομίζω ότι πράγματι είναι μια σημαντική προσπάθεια. Αναζητήθηκε και αναζητείται συμβιβαστική πρόταση. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει, αλλά θα ήθελα να την ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και τις δύο επιτροπές για το πάθος, αλλά και την αφοσίωση που επέδειξαν ε, σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει το θέμα της ε, ποιοτική εργασίας, αλλά επίσης ε, είναι και απαραίτητο να δημιουργηθούν οι βέλτιστες δυνατές συνθήκες, γιατί υπάρχει πράγματι πάθος, ευθεία, ποιότητα δουλειάς, όλα αυτά πρέπει να μπορούν να εκφράζονται πλήρως. Και υπάρχει ένα όραμα που είναι ότι θα πρέπει να αναδιεργοθούν πλήρως ε, τα ωράρια εργασίας ε, στις επιχειρήσεις. Εμείς ε, θα συνεχίσουμε να συγκρόμετα για όλα αυτά τα θέματα και θέλω να εκφράσω την ευχή μου ότι θα υπάρχει τελικά η θέληση όλων να ολοκληρωθεί μια δουλειά που είναι πολύ σημαντική και που αφορά όλες τις γυναίκες σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, Επόμενη, η κυρία Βυσνιέσκα, η οποία είναι σκιώδης συγγήτρια από την Επιτροπή για την Ισότητα των Δικαιωμάτων των Γυναικών. Δεν είναι όμως εδώ. Δεν είναι παρούσα στην αίθουσα. Μάλιστα. Να περάσουμε λοιπόν στην ε, σκιώδη της Άλντε, Αντζέλικα Μνινάρ. Ούτε αυτή. Η κυρία Κούνεβα από την Κούβα. Σκιώδε από την Κούα. Έχει το λόγο. we're here. Okay. Α, ήταν εδώ η εκπρόσωπο τη Άλτε. Εκπροσωπείτε λοιπόν την ομάδα της Άλτα. Πάρτε το λόγο παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σκιώδης ε, της Επιτροπής Απασχόλησης και όντως ε, πρέπει να σας πω ότι έχω καταθέσει μια σειρά τροπολογιών και από πλευρά των συναδέλφων από, τις, ε, από την Επιτροπή ΘΑΜ. Να ευχαριστήσω καταρχάς ε, τους εισηγητές, τις εισηγήτριες για τη δουλειά που έχουν κάνει έω τώρα σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Συμφωνώ δε με αυτά που μόλις ακούσαμε σε ό,τι αφορά τον τίτλο της έκθεσης. Εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων, αλλά πέραν τούτου θέλαμε να επικεντρωθούμε στην ισορροπία Επαγγελματική και ιδιωτική ζωής και ακόμα και στα αγγλικά. Το νόημα είναι αυτό. Μιλάμε για μια ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής ζωής και επαγγελματική ε, ζωής. Όπως σας είπα, από κοινού με τους συναδέλφους της ΑΛΔΕ, κατέθεσα μια σειρά τροπολογιών για ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι ουσιώδους σημασίας για την ομάδα μας. Καταρχάς, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο στην κοινωνία μας να υπάρχει πολιτισμική αλλαγή της νοοτροπίας σε ό,τι αφορά το ρόλο που διδραματίζουν τα φύλλα. Και αυτό πόσο μάλλον δεδομένου ότι υπάρχει και διαφορετική προσέγγιση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια κράτη-μέλη είναι πολύ πιο προοδευτικά. Και λόγω των δομών που υπάρχουν για τη φύλαξη και την ε, πρόνοια σε αυτές τις χώρες, αλλά και κάποια άλλα κράτη είναι σε πιο δύσχερη θέση. Δεν είναι μάλλον τα κράτη-μέλη αυτά που βρίσκονται σε δύσχερη θέση, αλλά οι γυναίκες των κρατών μελών αυτών, λόγω των περιορισμών που αντιμετωπίζουν έλλειψη πρόβλεψης για φύλαξη, ε, προβλήματα έλλειψη κινήτρων για την επάνωδο στον επαγγελματικό βίο. Θεωρώ ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να έχουν ευκαιρίες να μείνουν στο σπίτι παραπάνω, αλλά για να επανέλθουν στον επαγγελματικό στίβο. Εκ παραλλήλου είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι αυτό δεν είναι μόνο ρόλος του κράτους δεν επαφίεται μόνο στο κράτος να παρέχει τέτοιες καλύτερες δυνατότητες φύλαξης. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί μια κοινή προσέγγιση με όλους τους εμπλεκομένους φορείς και τους κοινωνικού εταίρους. Όχι μόνο να υπάρχει δηλαδή καινούργια νομοθεσία, να υπάρχουν και βέλτιστες πρακτικές, ανταλλαγή αυτών με άλλα κράτη-μέλη, να προσαρμόζονται αυτά στις εκάστοτε καταστάσεις που επικρατούν σε κάθε χώρα. Σημαντικό σκέλος είναι φυσικά η παράδοση και η προσέγγιση των γυναικών. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επιτρέπουμε να διανύζονται καταστάσεις όπου οι γυναίκες υπόκεινται διακριτική μεταχείριση. Αντιθέτως, θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια ευαισθητοποίησης για τα θέματα ίσης αντιμετώπισης και ίσων δικαιωμάτων και των ειδικών δικαιωμάτων που πρέπει να έχουν οι γυναίκες σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας. σε μια άλλη έκθεση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της οποίας είμαι εγώ εισηγήτρια, για την οδηγία μη διακριτικής μεταχείρισης στην αγορά εργασίας. Δεν ε, μας προκαλεί λοιπόν έκπληξη ότι πολλές από τις τροπολογίες είναι λίγο πολύ κοινέ με τις εκθέσεις αυτές. Είναι σημαντικό αυτό, ξέρετε, για να δοθεί και ένα συνεκτικό μήνυμα από πλευράς του Κοινοβουλίου προς τα έξω. Και Υπό την άποψη αυτή, θεωρούμε ότι η συλλογή και η αξιολόγηση αξιόπιστων ε, ομαδοποιημένων ε, ε, δεδομένων για το ρόλο των φίλων και την ισότητα και μάλιστα σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι σημαντικό και πάλι επαφίεται στους κοινωνικούς εταίρους και στους εμπλεκομένους φορείς να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά, τα δεδομένα αυτά και παράλληλα να παρέχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς καταγγελίας για όσους πλήττονται. Να καλωσορίσουμε την προσέγγιση του Προγράμματος Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2016, δεδομένου ιδιαίτερα του γεγονότος ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ισορροπία επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου, με σκοπό να αυξηθεί η συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Τέλος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα που παρέχει η ψηφιοποίηση. Γιατί η μεγαλύτερη αποδοτικότητα θα επιτρέψει και πιο προσαρμοστικές και ευέλικτες μορφές προσαρμογής του επαγγελματικού βίου λόγω ιδεολογίας, αν θέλετε. Κάποιες από τις ε, τροπολογίες που κατατέθηκαν από κάποιες πολιτικές ομάδες ενδεχομένως να μην συνάδουν και να μην συμπατίζουν με την απόψή μας. Είμαι ωστόσο πεπισμένη ότι μέσω των διαπραγματεύσεων στους κόλπους των συναντήσεων των σκιωδών τελικά θα καταλήξουμε σε συμφωνίες που τελικά θα αποβούν προς όφελος όσων πραγματικά χρειάζονται αυτή την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και δικού βίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Τώρα έχει το λόγο, κυρία Κούνεβα. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 4-6-4. Τόσο ήταν οι ανθρωπολογίε που κατατέθηκαν για την έκθεση αυτή. Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 751, όσο ο ρυθμός των Ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν και η έκθεση για την ισορροπία προσωπική και επαγγελματική ζωή, είναι στην αρμοδιότητα των Επιτροπών Employment και FAM αφορά όλες και όλους μας άσχετο επιτροπών κομματικών εθνικών ομάδων. διαβάζοντα κανεί τι τροπολογίε, θα δει πω το περιεχόμενο του τους φανερώνει τις μεγάλες αντιθέσεις που υπάρχουν όχι μόνο στα ίδια τα κράτη-μέλη τα οποία εφαρμόζουν διαφορετικές πολιτικές, αλλά και στο κοινοτικό μας δίκαιο που δεν έχει καταφέρει μέχρι το 2016 να ρυθμίσει και να εναρμονίσει ανοιχτά ζητήματα όπως την άδεια μητρότητας και την εικονική άδεια. Πολλές από τις 464 τροπολογίες, ίδιος αυτές που ήρθαν από τις δύο εισηγήτριες, την κυρία Μπλίνκεβιτσιούτε και την κυρία Σδάνοκα, που έκαναν εξαιρετική δουλειά, δίνουν ελπίδα για να προχωρήσουμε και να πιέσουμε πιο δυνατά ώστε να ξεκολλήσουν τα θέματα της άδεια μητρότητα, των γονικών αδειών, θέματα που έχουν τόσο φιλετική όσο και κοινωνική διάσταση. Δεν τα απορριθμίσω τις τροπολογίες αυτές να μας γλιτώσουν χρόνο. Έτσι και αλλιώς θα δουλέψουμε εντατικά για την σύνταξη των συμβαστικών τροπολογιών. Θα ήθελα όμως να σας θυμίσω τρία νούμερα. 8, 8, 8. Σας θυμίζω κάτι. Σας θυμίζει κάτι. Τότε επαναλαμβάνω. 8. Οκτώ ώρες δουλειά, οκτώ ώρες ελεύθερος χρόνος, οκτώ ώρες ύπνος. Ήταν το σύνθημα της εργατικής πρωτομαγιάς, διατυπωμένο ήδη από το 19ο αιώνα για να μας θυμίζει τις διαχρονικές αλήθειες. Κατά την ακρόαση που διοργανώθηκε το Μάη, η ομιλήτρια και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αποκαλύπτουν την καταστροφική επίδραση που έχουν οι συνθήκες εργασίας στην προσωπική ζωή και στην οικογένεια. Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι για να αξιολογηθεί ως ικανή, αποτελεσματική και χρήσιμη για την επιχείρηση και την υπηρεσία, δεν αρκεί να είναι έντιμοι, εργατικοί και μορφωμένοι. Πρέπει να είναι ευέλικτοι, ελαστικοί, ένα άνθρωπος λάστιχος, Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πολλοί από εσάς κατατέσατε τροπολογίες ζητώντας να διαγράφουν, να διαγραφούν ολόκληρες παραγράφοι ή αποδυναμώσατε παράγραφους, θεωρώντας πως δεν υπάρχει ανάγκη να ρυθμιστούν τα σημαντικά να ώστε να επιτευχθεί ισορροπία προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ναι, σε ορισμένες χώρες υπάρχουν ακόμη δικαιώματα και τηρούνται τα ωράρια. Είναι εξαιρέσει και όχι ο κανόνα. Το στρες, ο ανταγωνισμό στην εργασία, ο αγώνα για την προαγωγή σε κάτι κόστο, με κάτι κόστο, ο αγώνα για την επιβίωση των ανέργων, η παράταση των ωράριων και στο σπίτι μέσα το κομπιούτερ έχουν βάλει σε δεύτερη μοίρα την ίδια τη ζωή τελικά το ίδιο τον εργαζόμενο. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Να πιέσουμε και να αλλάξουμε τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ένωση. Να αλλάξουμε τις νομοθεσίες που αντί να επελευθερωθούν τους εργαζομένους, τους αφήνουν έρμια των πολιτικών και των κακών εργοδοτών. Εάν δεν θέλουμε να κάνουμε μια ακόμα έκτηση ιδιών έτσι, για να πούμε κάτι, πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη όθηση για την επανεκκίνηση των βελτιωμένων σχεδίων αναθεωρήσεις οδηγιών, αλλά να χαράξουμε από κοινό οι δύο επιτροπές το μονοπάτι που θέλουμε να, να δούμε την Ευρώπη να πηγαίνει. Και αυτό το μονοπάτι δεν μπορεί να είναι ο δρόμος της λιτότητας στη μητρική και εικονική άδεια, ώστε της ελαστικότητας συνεργασία. Ένα τέτοιο μονοπάτι οδηγεί μόνο σε αντίέξοδο. Ελπίζω με την σύνταξη συνεκτικών συμβαστικών τροπολογιών και με την υιοθέτηση προοδευτικών θεσίων <coughs> θα βάλουμε πλήρη, πλώρη για μια αληθινή κοινωνική Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Κούνεβα και τελευταία στο γύρο των σχεδόν εισηγητών ο κύριος Πιμέντα Λόπεθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την ανάλυση που κάνουμε της έκθεσης αυτής προκύπτει το σχόλιο ότι είναι απαραίτητη αυτή η ανάλυση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το συνδυασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Έτσι γενικά και αόριστα, αφηρημένα και αποσυνδεδεμένα από την πραγματικότητα. Και από τις βασικές αιτίες που είναι η αιτία των προβλημάτων που αναφέρονται και απαριθμούνται στην έκθεση. Θα πρέπει πρώτα να βρούμε τι αιτίε των προβλημάτων, γιατί τα προβλήματα έχουν συγκεκριμένε αιτίε. που οφείλονται σε μακροχρόνιες πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τις τελευταίες δεκαετίες είτε και λόγω επιβολής ή κατευθύνσεων καθοδήγησεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών τα βλέπουμε σήμερα. Αύξηση της φτώχειας, πάνω από 120 εκατομμύρια συμπολίτε μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 χωρών μελών βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχεια ή κάτω από το κατόφλι τη ένδυα. Ένταση των κοινωνικών ανισοτήτων, ένταση αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, αύξηση της επισφάλειας ή της έλλειψης ρύθμιση ε, στον χώρο εργασία, απαξίωση του, του μισθού και των εργασιακών συνθήκων των εργαζομένων. επίθεση κατά του κοινωνικού κράτους πρόνοιας και εξολόθρευση των κοινωνικών υπηρεσιών στις περισσότερες χώρες μέλη. Καταστροφή των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλειας, ασφάλισης, κοινωνικής προστασίας. Όλα αυτά τα μέσα, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί πρέπει να τα αποκρίνονται στις στοιχειώδεις ανάγκες των εργαζομένων ανδρών και γυναικών. Αυτά είναι τα προβλήματα και τις αιτίε τους θα πρέπει να εντοπίσουμε για να ξεκινήσουμε από τη διόρθωση των αιτιών πρώτα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ξεκινάμε από μια έννοια που κατοχυρώθηκε το 1919 με την δημιουργία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και ξεκινήσαμε από την έννοια της ισότιμης ε, ε, κατανομής μεταξύ εργασίας, ε, αναψυχής και ανάπαυλας. Και αφιερώνουμε 8 ώρες, κανονικά θα πρέπει να αφιερώνουμε 8 ώρες σε κάθε μία από αυτές τις πτυχές. Αλλά όχι μόνο δεν έχουμε γενικεύσει αυτή την πρακτική, το 8-8-8, 8 αλλά όλο και περισσότερο την υποβαθμίζουμε και απαξιώνουμε τους όρους ε, της καθημερινότητας και του βίου μας. Μπορούμε να μιλούμε για πολιτικές μητρότητας ε, και να τονίζουμε τη προσπάθεια υπεράσπισης της οικογένειας, στήριξης, προστασίας της οικογένειας, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτά χωρίς να, βρούμε, να αντιμετωπίζουμε τα αίτια του κακού. Επίσης, ε, έχουμε πολλές τροπολογίες που καταγγέλουν αφενός τις αιτίε, αλλά κυρίως δείχνουν το δρόμο για την αναβάθμιση των ε, ε, συνθήκων διαβίωσης που περνάνε από την αναβάθμιση των εργασιακών συνθήκων και την εξασφάλιση πρόσβασης στον πολιτισμό, στην αναψυχή, στον αθλητισμό και επίσης ε, θέτουμε ζητήματα αναβάθμισης ε, μισθολογικής, ε, αναβάθμισης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, βελτίωση των εργασιακών συνθήκων και στη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνεται αυτή η ανάγκη συνδυασμού και συμφιλίωση του προσωπικού και επαγγελματικού βίου. Επίση, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τι επισφαλεί θέσει απασχόληση και του υπερβολικά χαμηλού μισθού. Είναι αδύνατο να συνδυάσει κανεί την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή του αν ε, εργάζεται με βάρδιες ή εργάζεται κανείς τα Σαββατοκύριακα ή χρειάζεται να δουλεύει σε δύο δουλειές για να συντηρήσει την οικογένειά του. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και όλα αυτά τα θέματα. Η ρύθμιση του ωραρίου εργασίας επίσης είναι θεμελιώδους σημασίας. Και πέραν της ρύθμισης του οκτάωρου που θα πρέπει να είναι η ελάχιστη νομοθετική ρύθμιση, να μειώσουμε περαιτέρω το ωράριο εργασίας. Πριν από δύο μέρες, σε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΕΚΟΝ, ακούσαμε ένα επιχείρημα που δείχνει απόλυτη άγνοια ε, για τη μείωση του ωραρίου εργασίας στην Πορτογαλία στις 35 ώρες. Πρόκειται μια διαδικασία που δυστυχώς ισχύει μόνο στο δημόσιο. Και ήταν μια συνέπεια των μέτρων λιτότητας. Αλλά δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας χρησιμοποιήθηκε ε, για να στηριχθεί αυτό το επιχείρημα. Επίσης, το θέμα κοινωνικ και προστασία κοινωνικών παροχών, το ζήτημα τη γονική άδεια, άδεια, μεταποδοχών και μάλιστα πλήρων αποδοχών. Η ρύθμιση κάθε κράτο μέλο ε, είναι σημαντική, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, τι οδηγίες, τις εργασίες και να εφαρμόσουμε την οδηγία για τη γονική άδεια. Επίση, ε, δωρεάν δημόσιε υπηρεσίε για την παροχή φροντίδα. Ε, τους σταθμού, σταθμους η εξασφαλιση της πρόσβασης σε εκπαίδευση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ε, πλέον ε, δεν μπορείτε να μιλήσετε ο καθένας από σας πάνω από ένα λεπτό, γιατί έχουμε τέσσερις στον κατάλογό μας και μετά θα προχωρήσουμε με άλλο άλλη συνεδρίαση. Παρακαλώ. Η κυρία Κοσουόφσκα. Ε, Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τις συνεισηγητρίες γιατί α, πραγματεύονται ένα πολύ σημαντικό θέμα ανάπτυξης. Είναι σημαντικό ε, να συνδυάσουμε τον προσωπικό και, ή τον οικογενειακό και επαγγελματικό βίο γιατί μερικές φορές υπάρχουν αντιφάσεις και η πρόταση της Επιτροπής είναι περίπλοκη, ε, μη νομοθετική είναι σημαντικό ε, να κατοχυρώσουμε την ε, άδεια μητρότητας. Ε, το θέμα της ελαστικότητας, της πρόσληψης, της μορφής και της ευελιξίας. Σημαντικό για το συνδυασμό αυτών των δύο πτυχών. Αλλά επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη φροντίδα όχι μόνο των παιδιών αλλά και των ηλικιωμένων. Επίσης, πόσο μπορούμε, σε τι βαθμό μπορούμε τη μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία των ηλικιωμένων. Με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή την ανεξαρτησία των ηλικιωμένων. Ρομποτική, ιντερνετ, ψηφιακές τεχνολογίες ε, μας επιτρέπουν για ηλεκτρονική εκπαίδευση, τραπεζικές ε, εργασίες μέσω ηλεκτρονικού πάλι υπολογιστή, η ηλεκτρονική υγεία. Υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης ε, ανεξαρτησίας των ηλικιωμένων χάρη στις ε, ηλεκτρονικές αυτές τις ψηφιακές τεχνολογίες. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τον ψηφιακό αλφαβητισμό των ηλικιωμένων, ώστε να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία τους, γιατί όσο πιο απομονωμένοι είναι από το Ιντερνετ, τόσο πιο εξαρτημένοι θα είναι. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γεζοβιέσκα έχει το λόγο, Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τις ε, συνεισηγητρίες και από τις δύο γιατί είναι πολύ αξιόλογη η έκθεσή τους και χαίρομαι ιδιαίτερως που αναφέρθηκε η, η πρόσληψη με ελαστικέ μορφέ εργασία, γιατί πολύ συχνά στην Επιτροπή ακούω επικρίσει κατά αυτών των μορφών ελαστική εργασία η ευελιξία στην εργασία. Σε πολλέ χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτέ οι μορφέ εργασία, οι ελαστικέ εργασίε, δεν εξασφαλίζουν κοινωνική ασφάλιση. Οπότε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε αυτές τις μορφές, γιατί η ζωή μας έχει δείξει πόσο απαραίτητε είναι τέτοιες μορφές για την, για την κοινωνία μας. Βέβαια, θα πρέπει οι κυβερνήσεις να φροντίσουν ώστε και τέτοιες μορφές ευέλικτης εργασίας να καλύπτονται από κοινωνική ασφάλιση οι επιστήμονες ε, μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Στην Ευρώπη θα αντιμετωπίσουμε πραγματικό παλαιροϊκό κύμα, τσουνάμι με νέες μορφές απασχόλησης, ακόμη πιο ελαστικές, που σίγουρα δεν θα εξασφαλίζουν σταθερή ή πιο ασφαλή απασχόληση. Και για όλες αυτές τις νέες μορφές θα πρέπει να συζητήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να βρούμε λύσεις που θα βοηθήσουν τις κοινωνίες μας να υιοθετήσουν αυτές τις νέες μορφές που ούτως ή άλλως θα μας κατακλείσουν. Δεν μπορούμε να προστατευτούμε, δεν είμαστε απομονωμένο εσεί στην Ευρώπη. Υπάρχει αλληλεπίδραση και σύνδεση με τον υπόλοιπο οικονομικό κόσμο. Γι' αυτό ούτω ή άλλω δεν πρόκειται να αποφύγουμε αυτέ τι νέε μορφέ εργασία. Καλό θα ήταν λοιπόν να τι συζητήσουμε και να βρούμε κατάλληλε λύσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Σόιντροβα έχει το λόγο. Ε, ε, πρέπει να σας πω ότι είμαι ευγνώμων για την έκθεση αυτή και ξέρετε εγώ ε, δεν θα καταθέσω μόνη μου τροπολογίες γιατί εμείς ε, ως γονείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να συνδυάσει κανείς διάφορα πράγματα. Ένα μεγάλο κομμάτι της ε, ιδιωτική ζωής ε, έχει άμεση σχέση με την οικογενειακή ζωή. Επ' αυτού ελέγχθησαν πάρα πολλά και εγώ το βρίσκω πολύ καλό το γεγονός ότι συνεργάστηκαν οι δύο επιτροπές. Διότι Υπάρχει αυτή η σχέση με την ε, αγορά εργασίας, άρα δηλαδή αυτό το θέμα αφορά και τις δύο επιτροπές. Ε, υπάρχει και μια έκθεση σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων. Ε, εκεί προβλέπονται συγκεκριμένες διατάξεις για την αδιαμητρότητα, για το ευέλικτο ωράριο εργασία για τη γονική άδεια. Θέλω λοιπόν να επισημάνω ότι η φροντίδα των παιδιών είναι πλήρη απασχόληση. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αυτό όμω λείπει στην έκθεση. Εγώ πιστεύω ότι οι γονείς ε, πρέπει να μπορούν να απολάβουν καλύτερων προϋποθέσεων από άλλους απασχολούμενους. Μέχρι τώρα η φροντίδα των παιδιών ήταν κάτι που η κοινωνία δεν εκτιμούσε ιδιαίτερα, δεν του απέντε ιδιαίτερη σημασία. Ε, όσοι λοιπόν φροντίζουν παιδιά ε, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καλά τη δουλειά τους και ε, θα πρέπει να τους προσφέρουν και σχετικές θέσεις εργασίας γονική άδεια είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να ρυθμίζεται σωστά και στο έγγραφο εργασίας της ε, Επιτροπής προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πρέπει να τα εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Εμείς ως Κοινοβούλιο όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως πρόκληση και θέλω να πιστεύω ότι θα κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις και ε, σε αυτές θα συμβάλλουν και η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ και τελευταία η ομιλητριά μας, η κυρία Χέκ. Θα ήθελα και εγώ να σας παρουσιάσω την άποψη της Επιτροπής Γυναικών. Εγώ έχω καταθέσει ε, κάποιες τροπολογίες. Ε, θέλω να σας πω ότι για μας ε, είναι σημαντική η ισότητα των δύο φίλων. Πρέπει να επεκταθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ως βουλευτές φέρουμε ευθύνη. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει κοινωνία με ισότητα των δύο φύλων. Εμάς μας ενδιαφέρει ε, το πώς ε, μπορούν οι γυναίκες ε, να εργάζονται αργότερα, να συνταξιοδοτούνται. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανατροπεί η ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ούτε και να υπάρχουν επισφαλείς θέσεις εργασίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όταν μιλάμε για γονική άδεια, να ξέρουμε ότι από αυτού υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ε, σε ορισμένες ε, χώρες. Ε, οι γυναίκες είναι αναγκασμένες να μένουν στο σπίτι και να προσέχουν τα παιδιά είναι εγκλωβισμένες σε αυτή την κατάσταση και δεν έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν χρήματα. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν ε, ίδιες αμοιβέ ε, για ίδια εργασία. Από αυτού υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έχω καταθέσει και στατιστικά δεδομένα για να ξέρει κανείς που πρέπει να ξεκινήσει. Το όμως μας ενδιαφέρει να υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Ευχαριστούμε κυρία Χέντ. διαπιστώνουμε μετά από όλες αυτές τις παρεμβάσεις πόσο σημαντικό είναι το θέμα και πόσο ζωηρό ενδιαφέρον προκαλεί και στις δύο επιτροπές. Φαίνεται αυτό και από τον μεγάλο αριθμό των τροπολογιών. Γι' αυτό και εύχομαι καλή επιτυχία στις συνεισηγητρίες και στους και οδησηγητές προκειμένου να καταλήξουν σε συμβαστικές τροπολογίες ε, που θα εκφράζουν την κρατούσα άποψη και στις δύο επιτροπές και την επόμενη φορά στην κοινή μας συνεδρίαση θα ψηφίσουμε στις 12 Ιουλίου. Ωραία. Οπότε για να ολοκληρώσουμε αυτό το κοινότημα της συνεδρίασης Apple και ΦΑΜ να δώσω το λόγο στην συμπρόεδρό μου την κυρία Ουλσκοκ. Uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε αυτήν την αίθουσα θα συνεχίσουμε με την Επιτροπή Απασχόλησης που σημαίνει ότι καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ θα συνεργαστούμε η Επιτροπή Απασχόλησης και η Επιτροπή Γυναικών γιατί πραγματικά έχουμε κοινά θέματα, κοινέ υποχρεώσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα προχωράμε με την ε, κανονική συνεδρίαση της ε, Επιτροπής Απασχόλησης. Πάμε στο σημείο ε, υπαριθμών 15. Εκεί γίνεται λόγος για το άρθρο 33 προϋποθέσεις σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ε, και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στη Μάρθα Στίκινγκς από τον, Ευρωπαϊκό, από τον Φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Παρακαλώ, αν θέλετε μπορείτε να έρθετε εδώ, να καθίσετε στο Προεδρείο και μπορείτε να μας κάνετε μία σύντομη εισαγωγή σας καλωσορίζουμε. Ε, η συζήτηση θα γίνει μετά τη σύντομη εισαγωγή σας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Στίκινγκς.